Ε, διαβεβαιώσω ότι όλες οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Έχουμε ένα, μία πρόταση ψηφίσματος για να κλείσει η συζήτηση, η οποία τώρα έληξε. Η ψηφοφορία θα γίνει την 5η στις 11.30. Ευχαριστώ όλους και τώρα θα περάσουμε στις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού. ξεκινώντας από την κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Φεβρουάριο έπληξε ένα ανεμοστρόβλο στην Βίλα Ρεκόντε κάποιους παραγωγούς. Σε λίγα δευτερόλεπτα κατέστρεψε ο ενημεστρόβλος αυτό στην εργασία ε, μηνών για να μην πω ετών ε, θα πρέπει να αναδημιουργηθούν αυτές οι, οι εγκαταστάσεις τώρα. Στις 25 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους υπήρχε μια άλλη καταστροφή που επίσης κόστησε εκατομμύρια ε, ευρώ. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ για την τοπική ε, οικονομία. 2.000 ε, οικογένειες πλήττονται, 10.000 θέσεις απασχόλησης. Οι κλιματολογικές καταστροφές είναι όσο πάει και πιο ε, συνήθεις ε, πλήττουν την ε, <clears throat> δυνατότητα οικονομικής δραστηριότητας. τα ασφάλιστρα είναι πάντα τόσο ψηλά που δεν μπορούν να πληρώνονται από τους ενδιαφερομένους. Χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο ε, κατόφλι ε, ασφαλίσεων για όλους τους ε, παραγωγούς που θα βοηθούν από το Ταμείο Λεγγύης γιατί δεν θα μπορέσουν να ανασυγκροτηθούν ίσως βρεθούν στο περιθώριο λόγω των, της καταστροφής αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι όταν πήρατε το λόγο και μιλάτε περισσότερο από ό,τι προβλέπετε και μιλάτε πάρα πολύ γλίγορο που δεν μπορούν να μας εξυπηρέσουν γι' αυτό οι διερμηνείς. Παρακαλώ λοιπόν να είστε πιο σύντομοι, πιο περιορισμένοι. Η κύριε Σμόρκο. Σμόρκο, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ο Πρωθυπουργό Γιάνν φύγει ω ε, επίτροπο είχε έρθει στι Βρυξέλλε για να συζητήσει για τη μεταφορά οικονομικών πόρων από διάφορα τομεί, πρόκειται για 350 εκατομμύρια ευρώ όπως παιδεία και οικονομική ένταξη στον τομέα των μεταφορών. Χρειάζονται οι μεταφορές βέβαια αλλά έχουμε την στρατηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020 και σε αυτή την ε, ε, ε, περίοδο κρίσης θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση του οικονομικού κινδύνου προωθώντας την παιδεία. Αυτά έχουν την κύρια προτεραιότητα για τις οικονομίες. Συμφωνώ λοιπόν με τους ε, Σλοβάκους ε, δάσκαλους, εμπειρογνώμονες, πολίτες που δεν συμφωνούν με τις μεταφορές αυτές. Θα πρέπει να υποστηριχτεί η απασχόληση, η παιδεία. Πώς θα γίνει όμως αυτό, γιατί 350 εκατομμύρια ευρώ που πρόκειται να αφαιρεθούν είναι ένα τεράστιο, τεράστιο ποσό που θα κατασκευάσει την μία μόνο 11 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο ο κύριος Τρεμόσα Ιμπαλσέλς Ραμών. Αγαπητοί συνάδελφοι, τον περασμένο μήνα έκλεισε το τηλεοπτικό δίκτυο TV3 από την ε, ε, ε, κυβέρνηση αυτόνομης περιφέρειας. Αυτός ο αυτό το κλείσιμο ήταν ε, ε, παραβίαση των ε, οδηγιών ελεύθερης αναμετάδοσης αλλά ήταν επίσης και παραβίαση της αδελφοσύνης που ενώνει τους Καταλανούς και τους ε, κατοίκους της Βαλένθια από με μια κοινή γλώσσα επιβάλλονται κατο... κυρώσεις αξίας εκατομμυρίων ευρώ στους, ε, στην οργάνωση δράση για τη Βαλένθια και τους επιβάλλει μετά από χρόνια να κλείσουν τα τηλεοπτικά τους δίκτυα. Υπάρχει μια τοπική περιφερειακή πρωτοβουλία υπέρ της ε, τοπικής ε, καταλανικής τηλεόρασης η οποία παρουσιάστηκε ενώπιον του Ισπανικού Κοινοβουλίου με υπογραφές ε, άνω των 6.000 κατοίκων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λοιπόν αυτό από την κυβέρνηση, αλλά μέχρι τούτο δεν έχει γίνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Στρεμόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο υπόλοιπο μηχανισμό στήριξη στην ελλάδα ανακοίνωσαν πρόσφατα μια κυβερνητική δέσμευση για άντληση 50 δισεκατομμυρίων ευρώ από πώληση δημόσιας περιουσίας μέχρι το. 2015. Δηλώσει του εκπροσώπου της κομισιόν του κ. Ντερούζ εμφανίζουν ότι λέει πως το πραγματικό στίχημα της ελληνικής οικονομίας είναι η καθολική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας. η δημόσια όμως περιουσία στην ελλάδα δεν είναι όλη ίδια. άλλο είναι η εμπορική περιουσία όπως τα κτίρια που δεν επιτελούν δημόσιες λειτουργίες και άλλο μια βίαιη αλλαγή χρήσεων γης σε βάρος του περιβάλλοντος όπου απειλούνται ελεύθεροι χώροι όπως το πρώην αεροδρόμιο της αθήνας που προορίζονται να καλύψουν το έλλειμμα πρασίνου των μεγάλων πόλεων που διαθέτουν ανακάτοικο λιγότερο από τρία τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ενώ είναι δέκα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. απειλούνται και περιοχές κρίσιμης περιβαλλοντικής προστασίας όπως το δέλτα του νέστου όπου προκηρύχθηκαν ήδη τουριστικές εγκαταστάσεις χιλιάδων στρεμάτων. τέτοιες αλλαγές χρήσεων που θυσιάζουν ζωτικές περιβαλλοντικές λειτουργίες αποτελούν το αντίθετο κάθε ορισμού βιώσιμης ανάπτυξης. η κρίση και το χρέος δεν αναιρούν το δικαίωμα των επόμενων γενεών για ακέραιο φυσικό περιβάλλον και ευκαιρίες για βιώσιμες πόλεις. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Ο κύριος Μιγκάλσκι τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Κρίμα που ο κύριος Μακμίλαν Σκόλτ ε, σταμάτησε να προεδρεύει, διότι είχα ένα θέμα το οποίο θα τον ενδιέφερε. Ξέρω ότι τον ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχα λίγα πράγματα να πω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, μετά από τις εκλογές της 19 η Δεκεμβρίου, συγγνώμη, την παραμονή των εκλογών της 19ης Δεκεμβρίου στη Λευκορωσία, συνελήφθησαν αρκετά άτομα. Ένας εκ των συλληφθέντων, ο κύριος ε, Μιχαλέβιτς, απελευθερώθηκε στις 9 Ιανουαρίου και είπε ότι βασανίστηκε. Δεν θα σας κάνω την περιγραφή των βασανισμών που υπέστη, αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρό ο βασανισμός. αυτή την εβδομάδα ε, ε, θα υιοθετήσουμε ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, γι' αυτό και στρέφουμε προς την ε, Προεδρία, κυρίως τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Μακμίλαν Σκοτ, και του λέω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε σαφέστατα, δυνατά και καθαρά, ώστε να σταματήσουν αυτές οι απονείδησες πρακτικές. Ευχαριστούμε. Σας άκουσε ο κύριο Μακμίλαν Σκοτ ε, από την αίθουσα, βρίσκεται στα έδρανα, αλλά μας ενδιαφέρουν όλους τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν αναφέρεστε σε θέματα βασανισμών, σας διαβεβαιώ ότι ακόμα και ο Προεδρεύων αυτή τη στιγμή και του, τον έχουν βασανίσει και του έχουν βγάλει τα νύχια από τα δάχτυλά του ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ειδικά όταν μιλάμε για βασανισμούς και κάνετε λάθος αν λέτε ότι δεν μας ενδιαφέρουν βαθύτατα τα θέματα αυτά. Ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στις αρχές ε, του έτους υπήρχε στη χώρα μου ένα σύμνος ε, κατά της ε, προστασίας του περιβάλλοντος. Εμείς προετοιμάσαμε στο facebook μία διαμαρτυρία όπου καλούνται οι άνεργοι, εκείνοι που δεν έχουν δικαιώματα που έχουν ε, περιορισμένες εμβέλειας ε, ε, συμβόλαια εργασίας όλοι εκείνοι που στη χώρα μου δεν έχουν ωφεληθεί καθόλου από σπουδές τους που ζουν από 500 ευρώ τη ε, μήνα πάνω από 40.000 υπογραφές υπάρχουν στους ανθρώπους αυτούς στο facebook αυτή είναι η Ευρώπη μας αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να μιλήσουν για την τόσο δύσκολη θέση στην οποία ζουν, στην οποία ανασφάλεια. Οι άνθρωποι δεν έχουν δίκιο. Ευχαριστώ κύριε Πόρτας. Ο κύριος Αλαβράκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω για το θέμα Λιβύη. Η εξέγερση στη χώρα αυτή που ακολουθεί την Τινησία και την Αίγυπτο είναι πιο αιματηρή και εξελίσσεται δραματικά. εκ πρώτη όψεω οι λαϊκέ αντιδράσεις κατά του καθεστώτος είναι αυθόρμητες και ιδεολογικά αδέσποτε, στρέφονται εναντίον ενό καθεστώτος με προφανή αδυναμία να επιλύσει χρόνια προβλήματα ανάπτυξης και στοιχειώδους κοινωνικής δικαιοσύνης. η ευρώπη έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή κύριε πρόεδρε λιβύη δραστηριοποιούνται δεκάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρετανικές ιταλικές γαλλικές και πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ενώ η χώρα αυτή είναι τρίτη πετρελαιοπαραγωγός στην αφρική. η αστάθεια φοβίζει τις αγορές και ήδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει υπερβολικά. θεωρώ ότι υπό τις παρούσες συνθήκας η ευρώπη πρέπει ιδιαίτερα να προσέξει πρώτον τη διόγκωση του κύματος των προσφύγων όχι μόνο από τη λιβύη αλλά από όλη τη βόρεια αφρική και δεύτερον από την ανατροπή όλων των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών και την υπερδίνωση της οικονομικής κρίσης. επιπλέον κύριε πρόεδρε θα πρέπει να αξιολογηθούν τα αίτια και να λάβουμε μέτρα για το τι γίνεται μέσα στην ευρώπη ιδίως να δώσουμε δουλειά και προοπτική στους νέους διότι οι νέοι των χωρών του, του ισλαμικού τόξου δεν είχαν ελπίδα. γι' αυτό έκαναν αυτά τα οποία έκαναν και θα δούμε τι θα γίνει και εδώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Βαντίν Τουντόρ το λόγο τώρα. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες μέρες το κόμμα που έχει την κυβέρνηση στη χώρα μου, υιοθέτησε μία επονίδηση απόφαση, αποφάσισε να σκοτώσει, να θανατώσει όλα τα αδέσποτα σκυλιά. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους σοσιαλιστές της πολιτικής ομάδας των σοσιαλιστών να μην λερώσουν τα χέρια τους με το αίμα αυτών των αθώων σκυλιών. Ο Ιησούς Χριστός ε, αγαπούσε τα σκυλιά. Ίσως όλοι οι περισσότεροι έχετε σκυλιά στο σπίτι και το αγαπάτε σαν παιδί σας, αλλά η Ρουμανία επιστρέφει στο Μεσαίωνα, ξαναγίνεται βάρβαρη χώρα και περνάει στην ευθανασία των σκύλων που μπορεί να ε, αλλάξει και να οδηγηθεί και στην ευθυνεσία ανθρώπων. Βοηθήστε τη Ρουμανία να μην μετατραπεί στην Ουγγάντα του Ίνδια Μινταντά. Υπάρχουν ε, ειρηνικέ λύσεις, πολιτισμένε ε, λύσεις και το έγκλημα δεν έχει ποτέ λύσει τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Η κυρία Θεοχάρους έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι η προσοχή όλων μας στρέφεται τον τελευταίο καιρό στην εξέγερση των λαών της βορείου αφρικής ωστόσο δεν πρέπει να παροραθεί και η εξέγερση των τουρκοκυπρίων στην κατεχόμενη κύπρο είναι μια εξέγερση με ιδιαίτερη σημασία και ειδικά εκείνοι οι οποίοι κόπτονται ότι δεν ακούμε την φωνή των τουρκοκυπρίων αυτή τη στιγμή είναι η ώρα να ακούσουν πραγματικά την φωνή των τουρκοκυπρίων. οι τουρκοκύπροι έχουν εξεγερθεί εναντίον της οικονομικής δυσπραγίας που τους έχει επιβάλει η τουρκική κατοχή εναντίον της παρουσίας των επίκων οι οποίοι αλλοιώνουν τη σύνθεση του πληθυσμού και τους οδηγούν στην εξαφάνιση εναντίον της επέλασης του Ισλάμ με την ανέγερση εκατοντάδων τζαμιών και με τους θρησκευτικούς δασκάλους που στέλνει ο κύριος Ερτοάν στην κατεχόμενη Κύπρο και αγωνίζονται με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας για να επιβιώσουν οι τουρκοκύπροι έχουν πει όχι στο σχέδιο ανάν. δεν είναι αυτοί που ψήφισαν ναι υπέρ του σχεδίου ανάν το οποίο διχοτομούσε οριστικά την κύπρο. γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να ακούσουμε την εξέγερση των συμπατριωτών μου των τουρκοκυπρίων. σας ευχαριστώ πολύ. Gracias. Σας ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Ο κύριος Γιάννη δεν είναι στην αίθουσα. Να δώσουμε λοιπόν το ορολόγο στον κύριο Πυρίλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση της αλίας, του ερυθρού τόνου στην αλία, στη Μεσόγειο, εξακολουθεί να δημιουργεί ανυπολόγιστα προβλήματα στους αλίες η Ιταλική κυβέρνηση, ακολουθώντας τις αποφάσεις της ICAT, μείωσε τις ε, ποσοστώσεις αλίας ερυθρού τόνου μόνο για την επαγγελματική αλία τόνου. Ε, αυξήθηκαν οι ποσοστώσεις για την ε, αθλητική αλληλεία, μία απόφαση η οποία ζημιώνει τους αλληλείς, οι οποίοι ήδη βιώνουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Υπάρχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις και υπάρχουν ήδη προβλήματα γιατί υπήρχε παρέκκληση για την αλληλεία και του λευκού τόνου. Η Επίτροπος Δαμανάκη που είναι εδώ θα έπρεπε να ζητήσει το 2011 να επιτραπεί τουλάχιστον η αλληλεία του κυτρινότου ρερουτόνου στην περιοχή της Καλαβρίας με δυνατότητα και αναθεώρησης για το 2012. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πυρίλο. Η κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ τα όσα, ότι τα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή επέτρεψε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατανοήσουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αγνοούμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να καταγγείλω μια στη συμπεριφορά της κυβέρνησης της Ιταλίας που θέλει να διασώσει τον Περλουσκόνη από τις δίκες που μόλις ξεκινήσαν για πολύ σημαντικά παραπτώματα ε, και αδικήματα και αποπλάνηση ανηλίκου. Ζητούν από το ε, Συνταγματικό Δικαστήριο να αποφασίσει ποιο δικαστήριο θα πρέπει να δικάσει τον ε, κύριο Μπερλουσκόνη. Κατά πάσα πιθανότητα θα ζητηθεί δικαστή ad περσόνα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να αγνοούμε την την Ιταλική νομοθεσία και να κάνουμε παραβλέψεις ε, και να γίνονται όλες αυτές οι παραβιάσεις από πλευράς κ. Μπερλουσκόνη ο Ιταλικό λαό θα πρέπει να βοηθηθεί από το Ευρωκοινοβούλιο. Να σα πω και την εξή σύμπτωση. Ενώ ο κύριο Μπερλουσκόνη ε, επιτίθεται ουσιαστικά στη δικαιοσύνη, ο Υπουργό Δικαιοσύνη έρχεται να προσπίσει να συζητήσει και δεν, ε, στις Βρυξέλλες και δεν βρίσκει ούτε μία στιγμή για να μιλήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ίσως γιατί δεν θέλει να μιλήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφύγει τις ε, δύσκολε ερωτήσει που θα του θέσουν. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο, ήσασταν λίγο γρήγοροι και υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ζητά συγγνώμη πρόεδρος από τους διερμηνείς. Ήταν πολύ δύσκολο να διακόψω τη συνάδελφος η οποία είχε παρασυρθεί και εν τη μου τη λόγου μπορούσε και να σκοντάψει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Αλφάνο την επόμενη φορά να μιλάτε λίγο πιο αργά για να μπορούν να σας μεταφράζουν. Ο κύριος Βλάσακ τώρα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 236 της περισμένης εβδομάδα. Σύμφωνα με τον οποίο από την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτος δεν θα είναι πια δυνατό να γίνει η διάκριση για την ασφάλιση ε, βάση του φύλου. Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των ασφαλίσεων. Είναι τελείως παράλογο. Δηλαδή δίνει την εντύπωση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείε δεν επιτρέπεται να κάνουν μια διάκριση ανάλογα με το πόσο συχνά είχε ένα δυστύχημα αυτοκινηστικό ή κατά πόσο ένα σπίτι που βρίσκεται σε ένα βουνό απάνω κινδυνεύει από πλημμύρα. Γιατί είναι σαφές ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα από αυτοκινητικά δυστυχήματα μεταξύ των αρένων ε, και όχι των θύλων ενός πληθυσμού. Επίσης, άντρες έχουν ένα προσδόκιμο ζωής 73, οι γυναίκες 80. Αυτό λοιπόν είναι αντίθετο προς οποιασδήποτε ασφαλιστική θεωρία να δίνουμε την εντύπωση ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ άντρων και κοινωνικών για λόγους ασφάλειας. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Φερέιρα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, οι κοινωνικές συνέπειες τι εφαρμογή των λεγόμενων μέτρων λιτότητας επιδεινώνονται. Πολλοί συνεχίζουν να συσσωρεύουν τεράστια κέρδη, ενώ γίνεται η μη βιώσιμη ε, χρήση των εθνικών πόρων σε περιπτώσεις χωρών όπως η Πορτογαλία πρέπει να μην συνεχιστεί αυτή η πίεση που επιβάλλουν οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, επηρεάζονται μισθοί, αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης, αυξάνεται η επισφάλεια της απασχόλησης, η οικονομική διακυβέρνηση. Όλα αυτά θέλουν να τα επιβάλλουν στη θέληση του λαού. Η κατάσταση επιδεινώνεται στην Ευρώπη. Γι' αυτό αυτή η αυτή η οπισθοδρόμηση του πολιτισμού μας δεν είναι αναπόφευκτη. Κάποια άλλη κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρχει. Θέλουμε να στηρίξουμε όλες τις διαμαρτυρίες, τις απεργίες ε, και κυρίως ε, την απεργία που θα γίνει τις 19 του μήνα από τα συνδικάτα στην Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Η κυρία βέτμαν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι συνθήκες ζωής των Κυπρίων που ζουν στη Βόρεια Κύπρο είναι μη βιώσιμες, είναι απαράδεκτε. Παραδείγματο χάρη υπάρχουν συνεχεί παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τουρκία μεταφέρει πληθυσμό στην περιοχή αυτή της Κύπρου και είναι ω εκ τούτου υπεύθυνη για σοβαρή δημογραφική αλλαγή. Οι Τουρκοκύπροι ήδη έχουν γίνει μειονότητα στην πατρίδα τους και πολλά από τα ονόματα των χωριών έχουν αλλάξει. Δύο πράγματα έγιναν τι τελευταίε εβδομάδε. Η αντίδραση σε αντίδραση ε, τις διαμαρτυρίες του Ιανουαρίου υπέστησαν προσβολή από την Τουρκία, οι Τουρκοκύπροι. Θέλω κύριε Πρόεδρε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα πριν χαθεί ένα μέρος του ευρωπαϊκού εδάφους στην Τουρκία και να εξασφαλίσετε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΤΟΣ θα ε, ζει με ασφάλεια στην πατρίδα του. Ευχαριστώ την κυρία Βέρτμαν. Θα το μεταφέρουμε στον Πρόεδρο Μπούζεκ ε, το έτοιμά σας. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, πριν από λίγες ώρες ο οίκος αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε για μία ακόμα φορά την οικονομία της Ελλάδας. Προέρχομαι από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και πρέπει να σας πω ότι κάνουμε ισχυρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται για την οικονομία. Αλλά αυτή η απόφαση του οίκου Moody's είναι απολύτως αδικαιολόγητη. Γίνεται μόλις μία μέρα πριν από την δημοπρασία των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματείων δημοσίου πολύ κρίσιμο για την ελλάδα και λίγες μέρες πριν από τις κρίσιμες συναντήσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου στις 11 και στις 25 μαρτίου όπου θα ληφθούν πολύ σοβαρές αποφάσεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που υποφέρει από αυτές τις αυθαίρετες αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης. Είναι αναγκαία η ρύθμιση της λειτουργίας αυτών των οίκων αξιολόγησης και επειδή έχω το λόγο κύριε πρόεδρε θα ήθελα να πω και δύο κουβέντε για τα συμβούλια του μαρτίου. είναι πολύ κρίσιμο ο μήνα μάρτιο για την ευρωζώνη και για την ευρωπαϊκή ένωση συνολικά. μια αποτυχία θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ένωση. οι αγορέ θα κάνουν την αποτυχία πανολεθρία και πρέπει να το προλάβουμε. δεν υπάρχει χρόνο για καθυστέρηση. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ο κύριος Ιωάνν Έντσιου έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν συμφωνίε μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στη Ρουμανία, κυρίως στο ε, επιχειρησιακό τομεακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη. Στη Ρουμανία ο Πρωθυπουργό δεσμεύτηκε προσωπικώ να βελτιώσει τη χρήση των ταμείων αυτών. Δυστυχώ όμω τα αποτελέσματα ε, είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Οι ρουμανικές αρχές που διαχειρίζονται τα διορθωτικά ταμεία όχι μόνο δεν βοηθούν ε, όσους λαμβάνουν ε, επιδότηση από τα ταμεία, αλλά κάνουν ε, απεριόριστες ε, παραβάσεις και έως και εγκλήματα. Χρησιμοποιούνται, ιδιοποιούνται τους πόρους ε, και χρησιμοποιούν και πολλές φορές τα κονδύλια για πολιτικές δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει όσο το δυνατόν συντομότερο τις αρχές που διαχειρίζονται τα διαρθρωτικά ταμεία. Μόνο ο εξωτερικός δάκτυλος θα μπορούσε να σταματήσει τις καταχρήσεις που γίνονται σε μόνιμη βάση σε όλες τις δομές της εξουσίας στη Ρουμανία και ε, αποστερούν από όσους θα έπρεπε να λαμβάνουν επιδοτήσεις ε, ε, τα χρήματα αυτά. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πατεκόπ Γκάλαγκερ. Το Ταμείο στην Ιρλανδία από τότε που δημιουργήθηκε προσέφερε πάνω από 380 εκατομμύρια για χρηματοδότηση έργων και στη Βόρεια Ιρλανδία και στις περιοχές γύρω από τα σύνορα. Οι οικονομικά υποβεθμισμένες περιοχές έχουν πάρει 9,8 εκατομμύρια για τη στήριξη εκπαιδευτικών και κοινοτικών πρωτοβουλειών στην Ιρλανδία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον. Η... Αυτό συμπεριληφθεί στα πρόσφατα στα, κομμά... στα ταμεία και στα ποσά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι ε, δεν θα συμβεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει στήριξη παρότι είναι σημαντική η στήριξη αυτή, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν σε περιορισμένη και στοχευμένη βάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, την περασμένη ε, Κυριακή υπήρχαν ε, δημοτικές εκλογές ε, στην χώρα μου. Το κόμμα που εκπροσωπούσε την πολωνική μειονότητα είχε μεγάλες επιτυχίες. Και αυτό παρόλο το γεγονό ότι στην Ουκρανία τη χάνουν διακρίσεων εις βάρος τους οι Πολωνοί. Δυστυχώς δεν επιστρέφησαν τα εδέφα που έχασαν πριν από 50 χρόνια. Η δυνατότητα συμμετοχή στην παιδεία είναι περιορισμένη για τους Πολωνούς αυτούς. Ακόμα και τα ονόματα τους τροποποιούνται, δεν επιτρέπεται να τα γράφουν πολωνικά και ε, να αντιθέσει προς οπωσδήποτε ευρωπαϊκά πρότυπα και ε, των κανόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν επιτρέπεται να υπάρχουν και οι ονομασίες των πόλεων και των χωριών στα ε, πολωνικά. Θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριο Βίλι Μάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Δαμανάκη, θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μου είναι αντίθετη στην απόφαση που υιοθέτησε το Συμβούλιο Κατεπηγόντος για να παρατείνει για ένα χρόνο την αλληλευτική συμφωνία με το Βασίλειο του Μαρόκου. Είμαστε αντίθετοι διότι εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στη συμφωνία αυτή τα ύδατα της αυτόνομης περιοχής της Δυτικής Σαχάρας που όπως γνωρίζουμε είναι μία από τις ε, ε, λίγες περιοχές ε, της ε, Αφρικής που προστατεύονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Πρόκειται για ύδατα τα οποία δεν είναι του Μαρόκου, δεν είναι δικά τους ύδατα και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας ε, στην Συμφωνία. Υπάρχουν αποφάσεις διεθνών δικαστηριών και το Διεθνές Δίκαιο άλλωστε που αυτό ακριβώς ε, κάνει, προασπίζει τα δικαιώματα της περιοχής σε σχέση με το Μαρόκο. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν στη μελλοντική συμφωνία να μην περιλαμβάνονται οι Σαχαραούι στην ε, ε, συμφωνία με το Μαρόκο. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι στην απόφαση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει και η εμπειρία τώρα της Τινησίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί ως Ευρωπαϊκή Ένωση όταν παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τετσέιρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με το κανονισμό ΠΟΣΕΙ, προσεχώς. Αυτό είναι το πρόγραμμα που αφορά τις ακραίε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη νέα νομική κατάσταση μετά τη συνθήκη της Αβώνης και Επίσης ε, υπάρχει μια προσπάθεια να είμαστε πιο ευέλικτοι όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει τι περιοχέ αυτέ και γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί στο σημερινό σύστημα. Παραδείγματο χάρη, εδώ θα ήθελα να δώσω σαν παράδειγμα τη Μεδέρα. Θα πρέπει τα εμπόρια για τον ε, εισαγωγέ και τις εξαγωγέ ε, ξεχασμένων προϊόντων να καταργηθούν. Ε, επίσης αυτό ισχύει για προϊόντα γεωργίας, ε, αυτό ισχύει παραδείγματος χάνει για την παραγωγή μπανάνας. Απειλείται η καλλιέργεια αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμονισμένη εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να συμβάλλει και ο οργανισμός ΠΟΣΕΙ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Μπάρτεν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ενημερώσω για τις πρόσφατες εξελίξεις για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Πολλοί ε, εκδίδονται χωρίς πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του. Είναι αδύναμοι, δεν μπορούν να εξετάσουν τα δικαστήρια στοιχεία. Και τώρα υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Ο δόκτωρ Μιγέλ Νικουέλ, που είναι κάτοικος περιοχής μου αντιμετωπίζει πιθανότητα έκδοση στην Ισπανία, όχι για κάτι το οποίο έκανε, αλλά για ένα δίκημα που πιθανώς να αποφασίσει να διαπράξει στο μέλλον. Είναι κάτοικος Λονδίνου επί 20 ε, χρόνια και λόγω μιας επιθυμίας ενός ανακριτή κινδυνεύει να ε, ανατραπεί όλη η ζωή του. Όποιος ενδιαφέρεται, ευχαρίστω να τον ενημερώσω για την υπόθεση. Πότε θα αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο και θα συζητήσει τις αδικίες που γίνονται εξ στο όνομα μάλλον του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει στεναρή θάση για την ε, Λευκορωθία σύντομα. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ένα καθεστώς που επιτρέπει πολιτικούς κρατούμενους, δεν επιτρέπει την ελευθερία του τύπου και έχει λογοκρισία. Η δύναμη της Λουκασέγκο δεν είναι απεριόριστη. η δύναμη του Λουκασέγκο δεν είναι απεριόριστη και επομένως θα πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα να βγει από αυτό το απολετερχικό καθεστώς οι πρώην κομμουνιστικές χώρες έχουν πείρα από καθεστώτα σαν αυτό το οποίο ζει αυτή τη στιγμή η Λευκορωσία. Επομένως, βασιζόμαστε πλέον σε αρχές και αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παγώσει τα εισοδήματα του καθεστώτος Λουκασέγκο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επαφές μας με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κοινέ αξίες. Θα πρέπει να δώσουμε μια εναλλακτική λύση σε αυτή την κατάσταση, δεδομένου ότι μια χώρα με πολιτελεοχικό καθεστώ δεν έχει μέλλον στο ε, Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην κυρία Λεγκρίπ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ήθελα να περιοριστώ στο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας και σύγκλησης. Στις 11 Μαρτίου προβλέπεται η σύνοδος που γνωρίζετε και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένα τέτοιο σύμφωνο να εξεταστεί σοβαρά γιατί είναι πολύ σωστή ιδέα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς εννοούμε. Το σύμφωνο αυτό δεν είναι, τουλάχιστον για μένα δεν είναι, με τη μορφή που έχει τώρα, ένα ακόμη έγγραφο στον μεγάλο κατάλογο των ευσεβών πόθων που εκφράζονται εδώ μέσα, αλλά μία σοβαρή και επίσημη επιβεβαίωση του οικονομικού πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, δηλαδή περισσότερη σύγκληση μεταξύ των οικονομιών της Ευρωζώνης και μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική συνεργασία εφόσον είναι αναγκαίο οι χώρες μέλη να κάνουν μια προσπάθεια για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους διότι ο διεθνής ο παγκόσμιος καθιστά τελείως απαραίτητη την αύξηση αυτή της ανταγωνιστικότητάς μας και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο αγώνας κατά του δημοσίου χρέους, υπέρ της σταθεροποίησης του νομίσματός μας και γενικά υπέρ μεγαλύτερης οικονομικής, κοινωνικής και δημοσιονομικής ή φορολογικής σύγκλησης. Η διακυβερνητική μέθοδος έχει αποδείξει ότι δεν ε, έχει μεγάλη διαφορά από την ε, κοινοτική. Αυτά είναι στήρες συζητήσεις και όπως είπε και ο κύριος Ρόμπουης, πρέπει να καταλάβουμε ότι ή θα συνεννοηθούμε ή δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Αντιγκρίπο. Ο κύριος Σικέρσκι. Η θα συνεννοηθουμε η δεν προκειται να γινει τιποτα ευχαριστουμε κυριε αντιγκρυπο ο κυριος σικερσκι η ανταγωνιστικοτητα και το σύμφωνο αυτής είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για ποιο λόγο για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη και η εμπιστοσύνη σε αυτήν υπάρχουν πολύ χρήσιμες ρήτρες στο σύμφωνο αυτό μείωση του χρέους αναμόρφωση ή μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων αλλά εμπεριέχει και ορισμένους κινδύνους η πρωτοβουλία αυτή έγινε χωρίς, μεγάλες διαβουλεύσεις, χωρίς πολλές διαβουλεύσεις και αυτό δημιούργησε ορισμένες υποψίες ότι η Γαλλία και η Γερμανία θέλουν δήθεν να απομονωθούν και να τα κάνουν όλα μόνες τους. Ορισμένοι θεώρησαν ότι πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια να δημιουργηθεί Ευρώπη δύο ή και πολλών ταχυτήτων με έναν πολύ ανταγωνιστικό πυρήνα ενώ οι χώρες που δεν θα είναι στην Ευρωζώνη έχουν κληθεί με να συμμετάσχουν και αυτές αλλά αυτό είναι τακτική χειρονομία καθαρά. Το σύμφωνο αυτό πάντως θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρωζώνη σε απειλή για την ενιαία αγορά. Ευχαριστούμε κύριε Σικέρσκι. Λίγη εδώ αυτό το τμήμα. Είχαμε και την κυρία Ματέρα στο κατάλογο για τις μονόλεπτες, αλλά επειδή απουσίαζε